Dear President, Guten Abend, Καλησπέρα σας, συνάδελφοι. Άρχεται πάλι η συνεδρίαση και πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης είναι η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου για τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο κανονισμός για τη χρηματοδότησή τους. Η συγγήτρια παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο καλείται σήμερα να συζητήσει την ε, έκθεση την οποία εξεπώνησα υπ' ονόματι της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και αφορά στον κανονισμό που έχει σχέση με το ε, στατυ με το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων καθώς και τη χρηματοδότησή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογος κανονισμός, ωστόσο μέχρι στιγμής τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν απολαμβάνουν ενός καθεστώτος που είναι αντάξιο της συνθήκης της λισαβόνας και της ευρωπαϊκής ένωσης δηλαδή ένα καθεστώς όπως ορίζει το άρθρο 10 παράγραφος 4 της ε, συνθήκης της λισαβόνας το οποίο μιλά για τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της ευρώπης διότι δεν νοείται φυσικά πολιτικό ευρωπαϊκό κόμμα να λειτουργεί ως διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση ε, στο επίπεδο του βελγικού κράτους. Ε, γι' αυτό και πρώτον αποδεχόμενη την έκθεση του γενικού γραμματέα για τη χρηματοδότηση των κομμάτων αλλά και την εισήγησή του για τη δημιουργία καθεστώτος την εισήγηση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην προηγούμενη έκθεση του 2003 για την ανάγκη να υπάρξει καθεστώς αλλά τότε δεν είχε εγκριθεί ακόμα η συνθήκη της λισαβόνας ε, και τέλος την απόφαση του προεδρείου της 10 η Ιανουαρίου ε, η επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων μετά και από σοβαρή ακρόαση με όλα τα πολιτικά κόμματα τους προέδρους και τους γραμματείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και καθηγητές διακεκριμένους των οικονομικών και του συνταγματικού δικαίου καθώς και μετά από ακρόαση της διεθνούς διαφάνειας και ε, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου της ένωσης ενέκρινε αυτή την έκθεση στην οποία απαιτεί ζητά από την ευρωπαϊκή επιτροπή να φέρει αντίστοιχη πρόταση προκειμένου να υπάρξει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό καθεστώς πολιτικών κομμάτων. το καθεστώς αυτό βεβαίως θα έχει ορισμένα κριτήρια όπως ορίζει η έκθεση δηλαδή θα πρέπει να έχει σε τουλάχιστον 7 χώρες εθνικά κόμματα μέλη ή και περιφερειακά εφόσον οι περιφερειακές αρχές των χωρών αυτών έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες. Ε, ταυτόχρονα θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην αναγνώριση των ευρωπαϊκών κομμάτων και στη χρηματοδότησή τους. για να υπάρξει χρηματοδότηση θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εκλέξει τουλάχιστον ένα βουλευτή στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και βέβαια τα κόμματα θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν μέλη άτομα απλούς πολίτες ε, εκτός από το να έχουν κόμματα μέλη. αυτό βεβαίως ε, που προτείνεται ε, περιλαμβάνει όχι μόνο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αλλά και τα ιδρύματά τους. ζητείται λοιπόν και αυτό είναι το σημαντικό σημείο ένα νομικό πολιτικό και φορολογικό καθεστώς για τα κόμματα τα ευρωπαϊκά κόμματα στο πλαίσιο βεβαίως και υπό την ε, κάλυψη του ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος γενικότερα των ευρωπαϊκών νόμων. η επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων συζήτησε αρκετά το θέμα και κατέληξε σε αυτή την πρόταση με ελάχιστες διαφοροποιήσεις βέβαια που φαίνονται ε, μέσα στις τροπολογίες αλλά στην ουσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ε, πρόκειται για την ενίσχυση της δημοκρατίας πρόκειται για την ισχυρότερη παρουσία των πολιτών στο επίπεδο των ευρωπαϊκών οργάνων μέσω της δημιουργίας ενός τέτοιου καθεστώτος και βεβαίως στα θέματα της χρηματοδότησης ορίζεται ότι το 10% θα πρέπει να προέρχεται από ιδίους πόρους στα κόμματα ε, και ότι υπάρχει δυνατότητα ε, για τους δωρητές το 12.000 ευρώ που υπήρχε μέχρι σήμερα να γίνει 25.000. Ε, σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε ζητώ από την ολομέλεια φυσικά να υπερψηφίσει αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιαννάκου. Εκ μέρους της Επιτροπής, ο Επίτροπος ε, Σεφτσοβίτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία να συζητήσουμε την έκθεση για την, τα πολιτικά κόμματα και ευχαριστούμε την κυρία Γιαννάκου που συνέταξε αυτή την έκθεση πρωτοβουλία, διότι εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα παίζουν σημαντικό ρόλο για την οικοδόμηση της Ευρώπης συμμετέχουν και συμβάλλουν σε πολιτικά θέματα τα οποία εξετάζονται από την ευρωπαϊκή προοπτική πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφεύγοντας έτσι καταστάσεις όπου κυριαρχούν ε, εθνικά θέματα σε αυτές τις εκλογές. Κάτι που συμβαίνει, όπως ξέρουμε, πολύ συχνά. Χαιρετίζω λοιπόν τον πρωτοπόρο χαρακτήρα της έκθεσής σας και προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο μέλλον. Το άρθρο 12 του κανονισμού 2004-2003 ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2011 θα δημοσιεύσει έκθεση για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και τις ε, χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες και θα αναφέρει κατά περίπτωση τροπολογίε που πρέπει να γίνουν στο σύστημα χρηματοδότηση. Χαιρετίζουμε, όπω είπα, την έκθεση πρωτοβουλία τη κυρία Γιαννάκου και το ψήφισμα που τη συνοδεύει σαν θετικό βήμα. Αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η στοιχεία για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού και των χρηματοδοτημένων δραστηριοτήτων θα μπορούσε να βελτιωθεί και να είναι πιο ακριβές. Εν ώψη αυτών και ε, ε, ε καθώς επίκειται και η ψηφοφορία αύριο στο Κοινοβούλιο προσβλέπ, έχουμε σαν στόχο να συμπεριλάβουμε στη νέα νομοθεσία τον κανονισμό 2004-203. Όποτε θα χρειαστεί να υπάρξει νέος κανονισμός θα μελετήσουμε το θέμα και θα λάβουμε εφόσον χρειάζεται τις αναγκαίες πρωτοβουλίε. Η Επιτροπή σκέφτεται πόσο ο κανονισμός 2004-203 θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω μακροπρόθεσμα για να συμβάλλει στην ανάπτυξη πιο ισχυρών και πραγματικά υπερεθνικών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκά επίπεδο ώστε να δημιουργηθεί ένα πραγματικά ε, ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος. Γνωρίζω ότι δεν είναι πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο ζητεί να υπάρξει το σχετικό καθεστώς. Αυτό έγινε σε μία μελέτη και η οποία έδειξε σαφώς πόσο περίπλοκα συνταματικά και πρακτικά θέματα έχουν προκύψει για την ε, καθιέρωση ενός τέτοιου καθεστώτος. Είναι λοιπόν αυτό ένα θέμα που απαιτεί προσεκτική και ενδελεχή ανάλυση. Το ίδιο ισχύει και για κάποια άλλα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση προτάσεις που θα απαιτήσουν τροπολογία του χρηματοδοτικού κανονισμού, η Επιτροπή βλέπει την ανάγκη για ευρύτερη αντιμετώπιση του θέματος και πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά προτού καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα η έκθεση της κυρίας Διανάκου και το ψήφισμα που τη συνοδεύει οπωσδήποτε θέτει σημαντικά θέματα δημοκρατικού χαρακτήρα τα οποία χρειάζονται όλη την προσοχή μας και προσβλέπω στη συζήτηση που θα γίνει αυτό το θέμα απόψε και βεβαίως και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεύκοβιτς. Έχουμε λοιπόν εκ μέρους των πολιτικών ομάδων τον κύριο Κασίνη για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννάκου η οποία πραγματικά έκανε μια πάρα πολύ καλή και ευφύη δουλειά. Όταν μιλάμε για πολιτικά κόμματα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας δύο δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία είναι ότι σε καμία χώρα δεν ε, χαίρουν ιδιαίτερη εκτίμηση στα πολιτικά κόμματα. Και όταν γίνονται οι πολιτικές, ε, οι ευρωπαϊκές ε, εκλογές, όλοι θεωρούν ότι τα κόμματα τα εθνικά προάγουν τα δικά του συμφέροντα και όχι το ευρωπαϊκό συμφέρον. Έτσι λοιπόν, σε επίπεδο κοινή γνώμη δεν υπάρχει θετική στάση απέναντι στα κόμματα, αλλά ούτε απέναντι και στη λειτουργία τους προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να αντιδράσουμε όχι μόνο λόγω του συνθήκης Λιτσαβόνας αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπου η λειτουργία των κομμάτων κρίνεται εθνική, προστασία εθνικών συμφορών. Και αυτό δεν προάγει ούτε τη δημοκρατία, ούτε το κοινό καλό. Είναι λοιπόν να γνωρίζουμε ότι μιλάμε για το Σύνταγμα, ως εκ τούτου μιλάμε για ε, σημαντικά στοιχεία για το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε το κατσατικό των κομμάτων που είναι πραγματικά ευρωπαϊκά και δεν είναι απλά εθνικά μορφώματα τα οποία δεν έχουν μόνιμη δομή. Πρέπει να έχουμε κόμματα τα οποία πράγματι ε, θεωρούν αυτά ευρωπαϊκά ε, το καθήκον τους είναι πολύ μεγαλύτερο εάν πραγματικά θέλουμε να έχουμε και ένα ενιαίο ευρωπαϊκό εκλογικό νόμο ο οποίος ε, θα είναι πέρα από τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό λοιπόν θα βοηθήσει στο να αισθάνονται οι πολίτες ότι ανήκουν περισσότερο στην Ευρώπη. Ε, νομίζω ο κύριος Επίτροπος ανέφερε σημαντικότερα της δικής μου της παρέμβασης, αναφέρθηκε σε διάφορες ε, προτάσεις, αλλά υπάρχει ειδικά μία συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει ότι ε, θα πρέπει τα κόμματα να έχουν μια νέα νομική οντότητα που να ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη, να έχουν μια ενιαία οργανωτική μορφή και έτσι πράγματι θα εκπροσωπούν το ευρωπαϊκό κοινό συμφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γιαννάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υποσχέσεις σας ε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κύριο Κασίνη, επόμενος ομιλητής ο κύριος ε, Σάγκο δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Κύριε Γιαννάκη, να σας ευχαριστήσω για την κατάσταση που έχετε σε Πιστεύω ότι θα είναι πολύ και θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσμοθετήσει ένα καινούριο καλύτερο σύστημα που θα πλαισιώνει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ξέρετε, η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι όντως αντιπροσωπευτική το οικοδόμημα της αντιπροσωπευτική ε, δημοκρατίας έχει διατηρηθεί από τα μέσα... Ε, το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας έχει διατηρηθεί από τα μέσα του 19ου αιώνα μετά από τις ε, φιλελεύθερες επαναστάσεις έτσι ώστε ο λαός πλέον να πάρει την εξουσία στα χέρια του. Πιστεύω ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία βασίζεται σε πολύ γερά θεμέλια. Χρειάζεται όμως μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται νέους τρόπους για να εκφραστεί, με περισσότερη ποιότητα. Και νομίζω ότι το δικό μας κοινοβούλιο έχει κάνει πολύ καλή ε, δουλειά με την έγκριση αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν γίνεται, δεν νοείται δημοκρατία χωρίς ελεύθερη αντιπροσώπευση και δεν γίνεται να υπάρχει ελεύθερη αντιπροσώπευση χωρίς να υπάρχει ε, ελεύθερη συμμετοχή, πλουραλισμός στη δημοκρατία τα κόμματα, τα πολιτικά είναι αυτά που εκφράζουν το πλουραλισμό και είναι θεμελιώδη σημαντικά εργαλεία για την πολιτική εκπροσώπηση. Συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κοινή γνώμης, προσφέρουν εναλλακτικέ, προσφέρουν προγράμματα κυβέρνησης, διακυβέρνησης του τόπου και γενικότερης διακυβέρνησης αλλά και κατατομής. Ε, συντονίζουν τα κοινωνικά συμφέροντα, συμβάλλουν ε, στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ κυβερνώντων από τη μία και ε, των ετοιμάτων των λαών από την άλλη. Τα κόμματα δεν ε, δημιουργήθηκαν για να μάθουν στο λαό ποιες είναι οι ανάγκες των κυβερνώντων. Αντιθέτω, για να μάθουν στους κυβερνώντες ποιες είναι οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες των πολιτών. Αυτό είναι σαφές. Κάτι το οποίο λοιπόν έχει λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο, χρειάζεται τώρα να λειτουργήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να καθορίσουμε ένα πλαίσιο και να δώσουμε ευκαιρίες έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά πολιτικό πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις λειτουργίες που ήδη έχουν σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, θα πρέπει να έχουν ένα νομικό ε, καθεστώς στατή πολύ σημαντικό και αυτό προτείνεται με την έκθεση αυτή. Τα κόμματα που έχουν εδαφική παρουσία να ε, συμμορφούνται με τους δημοκρατικούς κανόνες επίσης. Ε, θα αναγνωρίζονται τα πολιτικά κόμματα και θα καθορίζεται η χρηματοδότησή τους ε, ενώ θα υπάρξει στήριξη από πλευράς κοινή γνώμης. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει μηχανισμούς και να διορθώσει τις ατέλειες του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, για δύο λεπτά ο η έκθεση της κυρίας Γιαννάκου ακολούθησε τη λογική των πρόσφατων εξελίξεων με σκοπό να αυξηθεί το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών. Για να ρυθμίσουμε το θέμα, η προσπάθεια να ρυθμίσουμε την κατάσταση των πολιτικών κομμάτων σημαίνει τη δημιουργία μιας κοινωνίας πολιτών χωρίς σύνορα. Αυτή η έκθεση είναι σημαντική επειδή θα ενισχύσει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ως προσωπικό όργανο της ε, Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 100 τροπολογίες προτάθηκαν για την έκθεση αυτό με 7 ε, ε, τροπολογίες ε, συμβιβασμού, κάτι που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Κοινοβούλιο για αυτή την έκθεση. Η ιδέα και, και η ιδέα να γίνει πιο, ευέλικτη, πιο, πιο ευέλικτο και πιο ελκυστικό το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης μεταξύ άλλων, ρυθμίζοντας μεταξύ άλλων το οικονομικό καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η ιδέα δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, αλλά να καθιερώσουμε ένα κοινό πρότυπο και να είμαστε βέβαιοι ότι τα κόμματα και τα ιδρύματα θα λειτουργούν με σύγχρονο τρόπο. Αυτή η έκθεση και οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να αλλάξουν το status, το quo στο οποίο, βάσει του οποίου τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αποτελούν μια προέκταση των εθνικών κομμάτων. Στα πλαίσια αυτής της φιλοδοξίας πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει δυνατότητα για, μεμονωμένα, ε, για μεμονωμένους πολίτες ε, να προσφορούν ως μέλη στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αναφέρθηκαν στην έκθεση ορισμένα ευαίσθητα θέματα. Γίνεται σωστά διάκριση ανάμεσα στο κριτήριο της ίδρυσης πολιτικού κόμματος αφενός και της χρηματοδότησής του αφετέρου. Η έκθεση πρέπει να υποστηριχθεί ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να δουλεύει πάνω σε ένα νέο κανονισμό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέφνερ, ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, το να υπάρχουν σαφείς κανόνες για τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη, ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να διαμορφώσουμε μια κοινωνία των πολιτών και για να προάγουμε τις πολιτικές συζητήσεις και για να υπάρχει η συμβολή σε αυτό το συνέστημα του ευρωπαϊκού, να υπάρχει ευρωπαϊκός προεκλογικός κανόνας με επιχειρήματα και οι κανόνες και οι εκστρατείες, με συγχωρείτε, να μην είναι εθνικές. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία για να ακούγεται την έκθεσή της. Εμείς ε, συμβάλαμε ουσιαστικά, δεν συμφωνούσαμε στην αρχή με όλα, αλλά με το αποτέλεσμα αυτό που προέκυψε είμαστε σαφώς ε, σύμφωνοι. Και θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία που για μας ήταν σημαντικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Παραδείγματος χάρη, εμείς πιστεύουμε ότι τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν ε, στον δημοκρατικό ανταγωνισμό πρέπει και αυτά να είναι δημοκρατικά. Και αυτό αφορά και κυρίως ε, τον καθορισμό των οργάνων, των ε, ληστών, των καταλόγων. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο υπερτιμών 5 και αυτό το βρίσκω μεγάλη πρόοδο. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που δεν θα τα αναφέρω, ε, θα αναφερθώ μόνο στα σημαντικότερα. Όσον αφορά το αίτημα ε, να υπάρχει ήδη ένας ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παλαιότερα προβλεπόταν ότι αυτό έπρεπε να ισχύει ε, για την αναγνώριση και τη χρηματοδότηση. Τώρα πια ισχύει μόνο για τη χρηματοδότηση. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να διαχωρίσουμε σαφώς την αναγνώριση από τη χρηματοδότηση. Αναγνώριση σημαίνει ότι μπορούν να υπάρχουν και νέα κόμματα με νέο πρόσωπο στην Ευρώπη. Αυτό δεν πρέπει να είναι περιοριστικό. Όσον αφορά όμως τη χρηματοδότηση, προφανώς ε, αυτήν μπορούμε να την συσχετίσουμε και με ένα ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας. Άρα δηλαδή εμείς συμφωνούμε με το αποτέλεσμα, έστω και αν θέλουμε να είναι λίγο πιο προβεβλημένο και γι' αυτό θα καταθέσουμε και μια τροπολογία. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Χέφνερ, επόμενος ομιλητής. Χέναν, Χάναν, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο ένα ψηφοδέλτιο που ρίχνουμε στην κάλπη κάθε τρεις και λίγο. Είναι, σημαίνει μια σύνδεση με, με την ε, κυβέρνηση. Δημοκρατία είναι ο Δήμος. Εμείς όλοι χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη και υπάρχει ο Δήμος το πρώτο συστατικό. Εάν αφήσουμε το λαό απ' έξω, μας μένει μόνο το κράτος. Δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει με γραφειοκρατικό τρόπο τους θεσμούς δημοκρατικής εκπροσώπησης. Είναι κάτι που προσπαθήσαμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε τις εκλογές, έχουμε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, έχουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά ε, κόμματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος νιώθει Ευρωπαίος. Ο κόσμος μπορεί να νιώθει ε, Ιταλός, Νορβηγός ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να θέλει να το βιώσει, να θέλει να βιώσει αυτή την ε, ταυτότητα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε χρηματοδοτώντας ή υπογράφοντας γραφειοκρατικά ένα σωρό χαρτιά. Εμείς Είμαστε κατά του ενιαίου καθεστώτος, είμαστε κατά των αυξήσεων του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό με, την, ε, με το τρέχον οικονομικό κλίμα και δεν ε, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, χρήματα για τις εκστρατείες αυτές. Δεν μπορεί κανείς να δημιουργήσει Ευρωπαίους δαπανώντας εθνικά χρήματα και εθνικά, αν θέλετε, κονδύλια, δημόσια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κύριο Χένεν για 1,5 λεπτό. Συνάδελφος κύριο Σούλτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ χαιρετίζω το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει σοβαρά το θέμα της υπόθεσης του εκδημοκρατισμού. Ο δρόμος βέβαια περνάει και μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των ε, ευρωπαϊκών κομμάτων, όπως το λέει και η κυρία Γιαννάκο. Ε, εδώ και κάποια χρόνια ε, τα κόμματα αυτά υπάρχουν, αλλά δεν αντιμετωπίζονται κάπως ισότιμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα ευρωπαϊκά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα ξεκινούν με παγίωσή τους, με αναγνώρισή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία τα κόμματα αυτά μπορούν να διερματίσουν σημαντικό ρόλο στις ευρωπαϊκές εκλογές, ε, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο επίσης στην κοινή γνώμη. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, εγώ θα ήθελα η εισηγήτρια να επιδείξει περισσότερο θάρρος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και μπορεί να κάνει ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Ένα βήμα το οποίο το αναμένουν πολλοί πολίτες και θα έπρεπε ίσως να γίνει. Θα έπρεπε να προβληθούν περισσότερο οι αποφάσεις σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα έπρεπε να προβάλλεται η κοινή δράση, η διαφάνεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει λοιπόν τώρα να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ προσβλέπω ε, σε μια επικοδομητική συνεργασία με τον Επίτροπο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σούλτς. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Άγνιου για ένα λεπτό. Η νομοθεσία αυτή θα σας επιτρέψει να ξοδεύετε χρήματα για τα εξασφαλίζοντας ότι θα αποκτήσετε το σωστό αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά θα γίνεται στην Ευρωμένο Βασίλεια ένα δημοψήφισμα κάθε φορά που θα προτείνετε κάποιες αλλαγές. Φοβάστε πάρα πολύ ότι μπορούμε να σας δώσουμε λάθος απαντήσεις. Σκοπεύετε λοιπόν να πάρετε από τους φορολογούμενους μας χρήματα για να τα καταθέσετε ε, για άλλους σκοπούς. Ο Άντρου Νταφ από τη δική μου περιοχή ευρωβουλευτής του οποίου το κόμμα κατέρευσε πρόσφατα και, διότι ε, αναζητώνται θεσμοί, θεσμικά όργανα, θεσμικά όργανα για να κυβερνούν το Ηνωμένο Βασίλειο σπέρνετε τους πόρους της δικής σας καταστροφής, διότι η νομοθεσία μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε εξτρατείες δημοψηφίσματος, κάτι που περιμένουμε εδώ και χρόνια στη χώρα μου. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να απομακρυνθούμε απόλυτα και πλήρως από τον έλεγχό σας. επιτρέπετε μία ερώτηση από τη κυρία Μάλιστα, η Σίνκλερ ε, θα υποβάλει την ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ο κύριος Σάγνου θα συμφωνούσε μαζί μου ότι ένα πολιτικό κόμμα που δέχεται χρηματοδότηση στα πλαίσια, σαν ενιαίο ευρωπαϊκό κόμμα θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις δραστηριότητες και, τις, και, τις, και το ρόλο του ε, ότι συμφωνούν δηλαδή με το, την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κινδυνεύει με τον τρόπο αυτό να χάσει τις αρχές του. Συμφωνείτε με αυτά κύριε Άγνου. Μου υποβάλλετε νομίζω μία ερώτηση, έτσι δεν είναι. Θα πάρουμε ό,τι μπορούμε, διότι εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει, θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του διαβόλου για να κάνουμε το έργο του Θεού. Παρέμβαση του κυρίου Σινκλέρ χωρίς μικρόφωνο, ακριβώς για αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Συνάδελφε Έγνιου, ε, κατά λάθο ε, σα αποκάλυψα Μπρόντ. Λάθο έκανα, με συγχωρείτε. Ήσασταν ο κύριο Γκρόντ, ο ε, συνάδελφο κύριο Μπρόντ ε, δεν ήρθε. Ε, γι' αυτό λοιπόν πάμε στον επόμενο μιλητή που είναι ο κύριος ε, Τρατσκόφσκι. Δύο λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννάκου και την Επιτροπή για τη θαυμάσια συνεργασία για αυτή την εξαιρετική έκθεση ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν Ευρωπαϊκό Δήμο, όπως μόλις είπε ο κ. Χάναν. Δεν το ξέρω αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκεί. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι να ενισχύσουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο ώστε να υπάρχει πιο ε, ζω... Ε, ζωηρή συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέματα και να πλησιάσουν περισσότερο στα θέματα που συζητούμε εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και τι το απλούστερο, να αρχίσουμε να συζητούμε ευρωπαϊκά θέματα ακριβώς με τους πολίτες. Και παρεπιπτόντος, δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, αλλά εγώ... Ε, δεν είμαι γραφειοκράτη, είμαι άμεσα εκλεγμένο μέλο αυτού του κοινοβουλίου. Σκοπό της συζήτηση είναι να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, στα οποία ανήκουμε όλοι. Ανεξάρτητα του γεγονότο αν καθόμαστε στην αριστερή, στο, κέντρο ή στην δεξιά πλευρά της αίθουσα, να βγούμε από τη σκιά, γιατί κανένα δεν ξέρει ακριβώ τι κάνουν τα κόμματα αυτά. Ποιο είναι το καθεστώς τους, προσφέρουν προστιθέμενη αξία ή όχι. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάποια προγράμματα και στο μέλλον να διεξάγονται για ευρωπαϊκά θέματα και ζητήματα ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς να καλύπτονται κάθε φορά από την εθνική ε, ρητορική. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα μα εξασφαλίσει κάποια ισορροπία ανάμεσα στι κοινοβουλευτικέ ομάδες σε άμεση σχέση με αυτά που συμβαίνουν εδώ στο Κοινοβούλιο, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερο, υπάρχει οργανωτική σύγκληση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα που είναι πραγματικά αξιέπαινα. Και τέταρτον, τρίτον, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, έχουν γίνει προσπάθειες που και αυτό νομίζω πρέπει να αποτελέσει στόχο όλων μας. Η κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δούμε την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη σύνθεση, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι είναι Ένωση κρατών μελών, αλλά είναι και μια πολιτική αρένα. Έχουμε πολύ μεγάλο δυναμικό και μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικά μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Υπάρχει ενιαία αγορά, ε, έχουμε ενιαία δικαστικά συστήματα σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, τα πολιτικά κόμματα έχουν τη δική τους ημερήσια διάταξη, αλλά και αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Με την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία, τη σταθερότητα στις κοινωνίες μας. Εγώ καλωσορίζω την πρόταση αυτή για την ε, τροποποίηση της χρηματοδότησης ε, των κομμάτων. Και θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για τη δουλειά της. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν ένα κοινό νομικό καθεστώς τα κόμματα αυτά. Είναι σημαντικό να γίνει αυτό. Και αυτό είναι εφικτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να το κάνουμε. Να εξετάσουμε και το εξής το δικαίωμα δημιουργίας Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος να δίδεται μόνο σε όσους φορείς ε, πληρούν συγκεκριμένους κανόνες. Π.χ. να διενεργούν ε, οικονομικούς ελέγχους, να σέβονται τις αρχές της διαφάνειας, να λειτουργούν σε ένα σωστά ρυθμισμένο περιβάλλον. Όλα αυτά είναι απαραίτητα και είναι προ όφελο του Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίο θα δει την καθημερινή του ζωή να βελτιώνεται ιδιαιτέρω. Το ενιαίο καθεστώ λοιπόν είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τα εμπρός. Μας βοηθάει στη σχέση μας με τους Ευρωπαίους πολίτες και προωθεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. κύριος Νταφ. Τα εθνικά, τα εθνικά, ε, πολιτικά κόμματα έχουν συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όμως, όχι τόσο όσο θα μπορούσαν. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα κενό, θα πρέπει να καλυφθεί και θα πρέπει εμείς να εργαστούμε περισσότερο έτσι ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη και να ε, συνειδητοποιήσει καλύτερα ε, τι ε, διαμείβεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Έχει έρθει η ώρα για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα οποία δεν θα αντικαταστήσουν βεβαίως τα εθνικά πολιτικά κόμματα, αλλά θα τα συμπληρώσουν. Θα μπουν στον πολιτικό στίβο για να αναζητήσουν τη στήριξη ε, των πολιτών προς τις ιδέες τους και προς τους υποψηφίους. Είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος σε όλη αυτή την αλυσίδα. Και είναι κάτι ε, που θα εξετάσει το Κοινοβούλιο το επόμενο μήνα και καλό τους πάντες να στηρίξουν την έκθεση της κυρίας Γιαννάκου προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με θάρρος και αισιοδοξία στην εμβάθυνση της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για ένα λεπτό, συνάδελφος Αλφονσί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η ίδρυση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ήταν ένα μεγάλο βήμα προς περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη. Εκφράζοντα τη βούληση των πολιτών της Ένωσης. Ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση η έκθεση Γεννάκου. Απλουστεύει και διευκολύνει την ίδρυση και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, περιορίζοντα την αντιπαροχή που θα απαιτηθεί για ε, δημόσιο χρηματοδότηση. Τα χρήματα θα αξιοποιούνται καλύτερα και θα θέλαμε τα ιδρύματα να έχουν δυνατότητα να λειτουργούν εκτό τη επικράτηση της όλα αυτά προωθούν ε, μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή δημοκρατία αλλά ο περιορισμό τη ελευθερία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων δεν θα ήταν η σωστή απόφαση. Ο κανονισμό θα απαιτεί μεταξύ των κριτηρίων αναγνώριση της ε, ε, πολιτικής εκπροσώπησης σε ένα κράτος μέλος να αποτελείται από εκπροσώπους του νομοθετικού σώματος ε, το δικό μας κόμμα ανοίξει στην Κορσική, μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό κόμμα εδώ και χρόνια, έχουμε συγκεντρώσει 26% των ψήφων στην Κορσική με πολλού μέλη στην συνέλευση. Επειδή δεν, δίνει στη συνέλευση της Κορσικής νομοθετικά δικαιώματα η Κορσική, δεν θα μπορούσε να υπολογιστεί. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή απόφαση και γι' αυτό ήθελα να επιστήσω σε αυτήν την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον ε, κύριο Αλφόνση. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ. Εσείς ε, πολύ αργά ε, σηκώσατε το, την μπλε κάρτα και δεν μπόρεσα να το δω. Δεν σας δίνω τώρα το λόγο. Λυπάμαι. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κιόρσκι, για ένα λεπτό. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να υφίστανται ε, για να έχουν ε, σωστές ρυθμίσεις να αποφεύγουν τις ε, καταχρήσεις. Οι υπερεθνικές δομές θα πρέπει να επηρεάζουν τα εθνικά κόμματα όμως δεν πρέπει να υπάρχει παρέμβαση ε, στα εσωτερικά μιας χώρας. Εγώ ως Πολωνός δεν μπορώ να δεχτώ μια κατάσταση όπου ένα πολιτικό κόμμα ε, μπορεί να ρυθμίζει τα της, ε, πολιτι... στη δική μου τη χώρα. Και επίσης οι φόβοι αυτοί υπάρχουν στους πολιτικούς και άλλων κομμάτων. Αυτό που θα πρέπει να υπάρχει θα πρέπει να είναι η χρηματοδότηση των κομμάτων γιατί σε εμά περικόπτεται τη η χρηματοδότηση και εμποδίζει ε, την ε, ε, πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κρατών, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προάγουμε τα κόμματα. Πρόεδρος διαδικαστικό, παρακαλώ συνάδελφε Βαντεστόκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είπατε πολύ σωστά ότι η δική μου η μπλε κάρτα ε, ήρθε πολύ αργά, δεν την είδατε, όμως δεν ισχύει αυτό. Ήδη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Νταφ ε, σας είπα ότι ε, θέλω να μιλήσω. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η διαδικασία. Μπορώ τώρα να σας δείξω την μπλε κάρτα ή θα συνεχίσετε τη συζήτηση. Γιατί εγώ έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Νταφ. Εκείνος μίλησε για διεθνικές λίστες ε, και έχω να κάνω μια ερώτηση από αυτού. Εντάξει, λέει ο πρόεδρο, αν θέλετε μπορείτε να την κάνετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να την υποβάλλετε. Λοιπόν, Πρόεδρε, το δικό μου το πρόβλημα σε αυτές τις διεθνικές λίστες του κυρίου Ντάφε είναι ότι εδώ έχουμε μια έκθεση για την οποία συζητάμε και το θέμα δεν είναι τόσο ότι υπάρχουν ε, ε, διεθνικές ε, λίστες. Εμένα αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι ότι εκεί προβλέπεται μόνο η συμμετοχή κομμάτων και εδώ γίνεται λόγος για κόμματα τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητα τουλάχιστον σε 7 χώρες. Το δικό μου όμως το κόμμα περιορίζεται μόνο στην Ολλανδία. Το τι κάνουν τα άλλα κόμματα μπορούν να κάνουν θέλουν, δεν μας διαφέρει καθόλου αλλά με αυτή τη ρύθμιση εσείς αποκλείετε κάποια κόμματα, ε, κάνετε λόγο για 25 έδρες. Μα πώς θα γίνουν όλα αυτά. Εμείς ε, λοιπόν θεωρούμε ότι μας αποκλείεται με όλα αυτά τα οποία προτείνετε. Συνάδελφε Στόπ ε, η ενδιάμεση ερώτηση είναι 30 δευτερόλεπτα και όχι η δική σας τοποθέτηση. Και άλλη φορά δεν θα σας ξαναδώσω και το λόγο. Η πρόταση που προωθώ είναι ένας υπερεθνικός διεθνικός κατάλογος από ένα τρίτο των κρατών μελών. Αν και ο κύριος Βαντεστόπ δεν μπορεί να προσελκύσει συναδέλφους με, που συμμερίζονται τις δικές του πολιτικές απόψεις από άλλες χώρες συνιστώ να εξετάσει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δικών του πολιτικών θέσεων. Ευχαριστούμε κύριε Ντάφ. κύριε κύριο για 1,5 λεπτό. Äh, Ευχαριστώ. På national plan, på europæisk plan og også på εγώ είμαι υποστηρικτή των πολιτικών κομμάτων ε, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Όμω με τα πολιτικά κόμματα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν μιλάμε μόνο για κομματικό μηχανισμό όταν μιλάμε για κόμμα. Μία από τι μεγάλε προκλήσει τη δημοκρατία σήμερα είναι ότι τα πολιτικά κόμματα εκφράζουν όλο και λιγότερο την κοινωνία. Είναι όλο και λιγότερο αντιπροσωπευτικά και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και ως εκ τούτου τα ευρωπαϊκά κόμματα χάνουν οπαδούς. Στη δική μας τη χώρα, στη Δανία, ε, πληρώσαμε, καταβάλαμε επιπρόσθετες ε, επιπρόσθετα κονδύλια στα κόμματα. Παρόλα αυτά όμως αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για τις ε, σχέσεις ανάμεσα στα νότατα στελέχη κόμματος και στη βάση. Τουν αντίον ελοχεύει ένας άλλος κίνδυνος, αυτός ο κομματικός μηχανισμός να αυτονομηθεί. Όσο λοιπόν περισσότερο αυτονομείται αυτός ο μηχανισμός από τους ε, οπαδούς, ε, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν είμαι επιφυλακτικός. Επιφυλακτικός απέναντι στην ιδέα του να υπάρχουν ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία θα χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια. Όχι γιατί είμαι κατά των κομμάτων, αλλά τα κόμματα θα πρέπει να σχηματίζονται από τη βάση, από κάτω προς τα πάνω να σχηματίζονται κόμματα. Και δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη αυτών των ευρωπαϊκών κομμάτων. Αυτός δεν είναι ο σωστό δρόμος για τη δημοκρατία, αλλά ούτε και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Επόμενο ομιλητή, ο κ. Αλαβράκος, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν συγχαίρω την εισηγήτρια κυρία Γιαννάκου για την ισορροπημένη και σωστή έκθεσή της και θεωρώ ότι η ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων με ευρωπαϊκή προοπτική που ξεπερνάει τα εθνικά σχήματα είναι καθοριστική για την κινητοποίηση της κοινή γνώμης στον χώρο της ένωσης και δημιουργία ενδιαφέροντος των πολιτών της ευρώπης να συμμετέχουν στα κοινά. διανύουμε κύριε Πρόεδρο, όπως είναι γνωστό μια εποχή απαξίωσης των πολιτικών αλλά και των πολιτικών κομμάτων στα οποία ανήκουν αφού οι ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν έρμεα των πολιτικών οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων. στην παρούσα λοιπόν συγκυρία η έκθεση της κυρίας γιαννάκου έρχεται να βελτιώσει την εμφάνιση των πολιτικών κομμάτων προς την κατεύθυνση ε, της ενοποίησης της ευρώπης σε μια αναγκαία μεταρρύθμιση που θα δημιουργήσει ευρώπη με ισότιμους πολίτες με κοινό πολιτικό νομικό και φορολογικό καθεστώς αλλά και ευκαιρίες ανάπτυξης. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαλαβράκο. Για ένα λεπτό η συνάδελφος κυρία Σινκλέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μίλησα προηγουμένως ε, για την εκλογική μου περιφέρεια, τα West Midlands και τις δυσκολίες που περνάνε. Δεν θέλουν ασφαλώς να ξοδεύονται περισσότερα χρήματα για τους πολιτικούς και υπάρχουν ήδη πολλοί ε, πολιτικοί που σπαταλάνε τα χρήματα του λαού θέλετε να δημιουργήσετε ακόμα ένα βήμα για, για να δημιουργήσετε το υπερ, ευρωπαϊκό υπερκράτος που θα συμπεριλαμβάνει και ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αυτό επιδιώκεται και οι πιο ευρωεσκεπτικιστές του Κοινοβουλίου είναι πρόθυμοι να πουλήσουν ε, τα, πιστεύω τους για να πετύχουν αυτό το σκοπό. Κάτι που το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο. Ευχαριστούμε κυρία Σινκλέρ. Για δύο λεπτά η κυρία Νεντέλτσεβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στις δημοκρατίες το κοινοβούλιο είναι η φωνή του λαού και υπάρχουν και τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματά τους που είναι εκείνοι που προωθούν ιδέες και δίνουν ζωή στη συζήτηση. Τα κοινοβούλια είναι η κινητήρια δύναμη των κοινοβουλίων και τα πολιτικά κόμματα τους δίνουν ουσία. Στο κοινοβούλιο μας ε, ε, ε, θρυνούμε διαρκώς για την έλλειψη ενδιαφέροντος του, των πολιτών για την Ευρώπη και την απουσία τους και από τα, τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η θέση που θα δώσουμε στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, στο δημόσιο χώρο που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Έχουμε κάνει πολλά με τη συνθήκη της Λισαβόνας και την πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Πρέπει τώρα να δώσουμε στα πολιτικά κόμματα τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες τους. Δεν νομίζω ότι τα μέσα αυτά όμως πρέπει να επιτρέψουν στα μεγάλα κόμματα να γίνουν, ε, να, να, να, να σκίσουν η ηγεμονία πάνω σε όλους. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να πείσουμε τους πολίτες ότι τα, Ευρωπα... τα πολιτικά κόμματα δεν είναι ε, ε, εγκαταλελειμμένοι της δημοκρατίας Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν δημόσιο ευρωπαϊκό χώρο που θα στηρίζεται σε σωστούς κανόνες χρηματοδότησης και στην διαφάνεια αυτής χρηματοδότησης. Δεν πρέπει να ευνοηθούν τα μεγάλα κόμματα σε βάρος των μικρών και αντίστροφα. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να, αναφερθεί, να αναφερθώ αφορά τη συνέχεια που θα εξασφαλιστεί ανάμεσα στο εθνικό, το ε, ε, περιφερειακό και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό καθεστώς πρέπει να, ε, να συνάδει με τις εθνικές νομοθεσίες ώστε όλα τα επίπεδα να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και πρέπει να δούμε και από πολύ κοντά αυτά που αναφέρεται στην παράγραφο 23 της έκθεσης κατά πέκτηση πρέπει να σκεφτούμε στο δεσμό που τα ευρωπαϊκά κόμματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν με εκείνα των άλλων περιοχών του κόσμου. Οι δημοκρατικέ αξίε που πρεσβεύουμε πρέπει να τι μοιραστούμε με του εταίρου μα στι υπόλοιπε περιοχέ του πλανήτη. Διότι σε μια, στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που ζούμε σήμερα, πρέπει εκείνοι που λαμβάνουν τι αποφάσει να προτείνουν από κοινού λύσει στα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντελέτσεβα. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Μπαλκιτσής. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και αυτό έχει υπογραμμιστεί στη συνθήκη της Λισαβόνας ώστε να υλοποιηθεί ο ευρωπαϊκός δημόσιος χώρος. Δουλειά μας είναι να ενθαρρύνουμε τους πολίτες, να ενδιαφερθούν περισσότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Χρειαζόμαστε διαφάνεια, σαφούς, σαφείς κανόνες στη λειτουργία των κομμάτων αυτών. Θα πρέπει να έχουν ίσο ε, καθεστώς νομικό αλλά και ε, χρηματοδοτικό, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να καταλάβουν πολύ καλά πώς λειτουργούν τα κόμματα αυτά. Θα πρέπει να διοργανώνονται τα κόμματα αυτά εσωτερικά, με σωστές αρχές, επάνω σε σωστές αρχές και να γίνεται πάντοτε σεβαστός ο κανόνας της διαφάνειας. Ευχαριστούμε ο κύριος Τάιν, η Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα ευρωπαϊκά ιδρύματα είναι εκείνα που έχουν συσταθεί ε, κυρίως με βελγικό δίκαιο. Αυτά τα ευρωπαϊκά κόμματα τι κάνουν ακριβώς. Συζητούν για ευρωπαϊκά θέματα, διοργανώνουν ε, συνέδρια και ε, είναι απαραίτητα για να μεταρρυθμιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα πρέπει να βοηθήσουν να υπάρξει ευρωπαϊκή δημοκρατία, ένα πολιτικό χώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αύριο λοιπόν θα έχουμε την έκθεση πρωτοβουλία ε, για να ψηφιστεί και η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύτερα να μεταρρυθμίσει τα κόμματα αυτά. Στο μέλλον θα έχουν ευρωπαϊκή νομική οντότητα. Οι φιλελεύθεροι εμεί θέλουμε να υπάρχει σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην αναγνώριση των κομμάτων και ε, στη χρηματοδότησή τους. Ε, αυτό που επίσης έχει σημασία είναι τα ευρωπαϊκά κόμματα να είναι δημοκρατικά, κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, ε, κυρία Τάιν, έχουμε τώρα τον συνάδελφο Βαν Όρντεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, ε, τα πράγματα πάνε προς μία κατεύθυνση και πολύ συχνά το Κοινοβούλιο πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν ζητούν ε, διεθνικές ε, λίστες. Τώρα θέλει το Κοινοβούλιο μας να σπαταλήσει περισσότερα εθνικά κονδύλια ή κρατικά κονδύλια. Μιλώ με την ιδιότητά μου του Προέδρου της, του New Direction, ενός φορέα για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση. Είναι απαράδεκτο να αυξάνεται το κόστος με τόσο γρήγορο ε, ρυθμό. Το 2009 6,9 εκατομμύρια ευρώ εξοδεύτηκαν. Το 2012 θα φτάσουμε στα 12,3 εκατομμύρια ευρώ, το διπλάσιο. Κάποιοι λένε αφού είστε κατά γιατί το Ίδρυμά σας δέχεται χρηματοδότηση. Απαντούμε εμείς διότι και λέμε το εξής, εάν δεν δεχθούμε τα κονδύλια αυτά θα διανεμηθούν στους άλλους, στις άλλες πολιτικές ομάδες. Ουσιαστικά έτσι αν αρνηθούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδοτούμε τις ε, δραστηριότητες των πολιτικών μας αντιπάλων. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιστραφούν χρήματα ε, στα εθνικά θησαυροφυλάκια. Ευχαριστώ. Κύριε Σκούντης, παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτό από την οικονομική κρίση δοκιμάζεται από κρίση δημοκρατία και κρίση νομιμοποίηση. Οι που εφαρμόζονται εξοργίζουν και απογοητεύουν τους πολίτες οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων τους απομακρύνουν από τη συμμετοχή όπως έδειξαν οι πρόσφατες ευρωεκλογές. γι' αυτό κάτω από προϋποθέσεις τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με τα ιδιαίτερα πολιτικά τους χαρακτηριστικά μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των πολιτών στη διεκδίκηση λύσεων υπέρ των λαών και όχι των οικονομικά ισχυρών οι κανόνε λοιπόν πολιτική και νομική αναγνώριση και η αναγκαία χρηματοδότηση πρέπει να διευκολύνει τη δράση του να αναπτύσσουν ελεύθερα τι πολιτικέ του τι εναλλακτικέ του προτάσει αυτή είναι η ουσία τη δημοκρατία και να είναι ανεπηρέαστοι από εξωτερικού περιορισμού πολιτικού ή οικονομικού. γι' αυτό έχω επιφυλάξει σε συγκεκριμένα σημεία τη έκθεση στο μέτρο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ω περιορισμή στην ελεύθερη και ανεξάρτητη οργάνωση και δράση των πολιτικών κομμάτων. η λειτουργία η δράση η οργάνωση των κομμάτων πρέπει να είναι θέμα δική του επιλογή και όχι κάτω από την αίρεση πολιτικού κυρίαρχου συσχετισμού. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή για την εφαρμογή του κανονισμού για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνει υπόψη την εμπειρία που υπάρχει από την εφαρμογή του κανονισμού σε οργανισμούς με ευρωπαϊκή προπτική. Η κυρία Γιαννάκου αποφάσισε να διατυπώσει κάποιες προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση του ισχύοντος νομικού περιβάλλοντος. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η πρόταση μετάβασης από το ισοδύναμο των βελγικών σε ένα ενιαίο νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Μια άλλη αλλαγή είναι η μεταβολή του ποσοστού χρηματοδότησης από ανεξάρτητες πηγές στο 10%. Το 2012 τα ευρωπαϊκά ιδρύματα και τα κόμματα θα πάρουν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μέγιστη διαφάνεια στη διαχείριση αυτών των πόρων. Προκειμένου να βελτιωθεί το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτέ τι αλλαγέ. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό. Συνάδελφο Βάντερ Στόπ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το κόμμα Party for Freedom ουσιαστικά ε, μιλάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των ε, συμφερόντων των κάτω χωρών. Εμείς δεν είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουμε όμως να ε, περιοριστεί στην οικονομική συνεργασία. Η εξουσία θα πρέπει να παραμένει σε κρατικό, εθνικό επίπεδο, διότι μόνο τα, σε εθνικό επίπεδο είναι γνωστό τι είναι, το, τι είναι το καλύτερο για τον εκάστοτε πολίτη. Στη συνθήκη της Λισαβόνας λέγεται ότι ορίζεται ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής συνείδησης και στην έκφραση, ε, στην προάσπιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω ότι είναι ε, γελία η δήλωση αυτή και απολύτως κατακριτέα. Το 2010 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να επιχορηγηθούν ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ουσιαστικά σπαταλήθηκε το χρήμα του φορολογούμενου. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί χωρίς τέτοιου είδους επιχορηγήσεις και θα πρέπει να καταργήσουμε τη διάταξη αυτή. Πολύ ωραία. Ο συνάλφο κύριο Τούσα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Το κεντρικό ζήτημα που βάζει η έκθεση για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων του είναι η δημιουργία ενιαίου καθεστώτος για τα ευρωπαϊκά κόμματα σύμφωνα με την ευρωενωσιακή νομοθεσία. η ευρωπαϊκή ένωση με την νομοθεσία της να καθορίζει ενιαίο τρόπο δομής και λειτουργίας για τα ευρωπαϊκά κόμματα να αναμειγνύεται στην εσωτερική λειτουργία τους στο καταστατικό και το πολιτικό τους πρόγραμμα. με πρόσχημα την δίθεν χαλάρωση του χρηματοδοτικού καθεστώτος ανοίγει το κουτί της πανδώρας με οικονομικές και κατ' επέκταση πολιτικές κυρώσεις σε βάρος των πολιτικών κομμάτων δηλαδή ασφιχτικότερο έλεγχο της λειτουργίας και της δράσης τους από την ευρωπαϊκή ένωση άσκηση πίεσης στα εθνικά πολιτικά κόμματα για βαθύτερη ενσωμάτωσή τους στην αντιλαϊκή πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης επίθεση στα κόμματα εκείνα που αμφισβητούν την αντιλαϊκή πολιτική τη στρατηγική της ευρωπαϊκής ένωσης την εξουσία του κεφαλαίου. δεν πρόκειται επομένως για κανένα κοινοβουλευτικό συντονισμό αλλά για ευρωπαϊκά κόμματα μηχανισμούς ιδεολογικούς και πολιτικούς της ευρωπαϊκής ένωσης για τη χειραγώγηση του εργατικού λαϊκού για αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε την έκθεση πρόταση για τα ευρωπαϊκά κόμματα τα πολιτικά ιδρύματα και τη χρηματοδότησή τους. Ευχαριστούμε κύριε Τούσα. Ε, πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και δίνω το λόγο στην κυρία Μπασέσκου. η διαφανής χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων είναι σημαντική για την υποστήριξη των δημοκρατικών αρχών. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό χώρο στον οποίο τα πολιτικά κόμματα θα αναλαμβάνουν δράση και οι πολίτες θα αισθάνονται ότι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους. Η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού, του ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος είναι ένα βήμα προς τα μπρος για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των κομμάτων. Έχουμε ένα νόμο του 2006 που άρχισε να εφαρμόζεται το 2010 και στο δημόσιο χώρο γίνονται συζητήσεις για τη χρηματοδότηση των υποψηφίων για την τοπική ε, αυτοδιοίκηση και το κοινοβούλιο που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα δημόσια κονδύλια. Το ανώτατο όριο είναι 1.600 ευρώ για κάθε υποψήφιο. Με τη χρηματοδότηση αυτή με, την εφαρμογή μεθέτας χρηματοδότησης θα, ε, θα εξαφανιζόταν η διαφθορά και θα μπορούσαμε να έχουμε αντί επαγγελματίες πραγματικούς υποψήφιους πολιτικούς. Η κυρία Ντότ ζήτησε το λόγο. Thank you, uh, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή απόψε δείχνει χαρακτηριστικά ποιο είναι το λάθος με την ευρωπαϊκή ατζέντα. Με μεγάλη έκπληξη άκουσα τα λόγια των προηγούμενων ομιλητών και με μεγάλη έκπληξη βλέπω για άλλη μια φορά πόσο μακριά είναι τα θέματα που συζητάμε εμείς από τον Ευρωπαίο πολίτη. Σωστά λέει ο κύριος Ντάφ ότι πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ ΕΕ και Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να το γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, αλλά δεν θα το καταφέρουμε με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ίσως θα πρέπει όντως να έχουν τους πόρους ώστε να καλύπτουν τις φιλοδοξίες τους τα πολιτικά αυτά κόμματα. Καλό τον κύριο Τάφ να πάει στην εκλογική του περιφέρεια και να πείσει και να τον πάρουν στα σοβαρά ότι όντως ε, έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Να δει πόσες, ε, πόσες ε, κοινωνικές ομάδες έχουν πληγεί ιδιαιτέρως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε τη Λισαβόνα, τον ε, αυξανόμενη ομοσπονδιακή Ευρώπη, η γραφειοκρατία, ε, τέτοιου είδους ε, θεσμικά όργανα, να δω αν θα πείσει τους ψηφοφόρους. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσει τη συζήτηση, ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω τις καταληκτικές παρατηρήσεις μου συγχαίροντας και πάλι την κυρία Γιαννάκου για την έκθεσή της διότι νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έδειξε σαφώς ε, πόσο σημαντικό, πόσο ενδιαφέρον υπάρχει το θέμα που έθεσε που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ανταλλαγή απόψεων έδειξε σαφώς επίσης πόσο ευαίσθητα είναι όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι αύριο το Σώμα θα εγκρίνει αυτή την πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρήσει τις υποχρεώσεις και θα ανταποκριθεί σε αυτό το ψήφισμα. Αλλά όπως είδατε στη διάρκεια της συζήτησης αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα θα απαιτηθεί δύσκολη και ευαίσθητη πολιτική δουλειά, διότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία από νομική και πολιτική άποψη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Η πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει σε ό,τι αφορά το καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Αλλά θα χρειαστεί να μελετήσουμε τη νομική βάση, το, νομικό σχήμα με ιδιαίτερη προσοχή και πιθανότατα θα χρειαστούμε διαφορετικά νομοθετικά κείμενα διότι η αναθεώρηση του κανονισμού 2004-2003 δεν θα επαρκεί διότι αφορούσε καθαρά το θέμα της χρηματοδότησης και όχι το θέμα του καθεστώτος των πολιτικών κομμάτων. Αυτή λοιπόν είναι μια οπτική γωνία στην οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Το θέμα που έθεσαν πολλοί ομιλητέ αφορά το, το τροποποίηση του χρηματοδοτικού κανονισμού. Και εδώ πρέπει να εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις ανάγκες και τα χρονικά περιθώρια και να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτά που αναφέρονται για μεγαλύτερη ευελιξία στην έκθεση. Το 2007 έγιναν κάποιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και θα εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις προτάσεις. Πρέπει ωστόσο να καταθήσω απόλυτα σαφές ότι δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για αλλαγές και να τις εντάξουμε όλες στην τρέχουσα διαδικασία αναθεώρησης του χρηματοδοτικού κανονισμού. Το Κοινοβούλιο είναι νομοθετικό σώμα και έχει τη δυνατότητα να θέσει το θέμα στην διοργανική διαδικασία εφόσον το επιθυμεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και προσβλέπουμε στη συνέχιση τη συζήτηση για αυτό το θέμα όταν ψηφιστεί το ψήφισμα και είναι και έτοιμη η απάντηση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο και για να ολοκληρώσει η συζήτηση η εισηγήτρια κυρία Γιαννάκο έχει το λόγο. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ε, Επίτροπο ε, για όσα είπε και για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε καθώς και τους συναδέλφους οι οποίοι στήριξαν την έκθεση αυτή νομίζω ότι έχει σημασία να επαναλάβω ότι όσο αφορά στη διαδικασία χρηματοδότησης τα κόμματα δεν ζητούν περισσότερα χρήματα και από την τροποποίηση του κανονισμού του 2007 έχει προκύψει μεγαλύτερη διαφάνεια όπως παραδέχτηκε η ίδια η διεθνής διαφάνεια. δεύτερον τα κόμματα είναι θεμητό να ζητούν ένα στάτους ευρωπαϊκό και την ευθυγράμμιση του καθεστώτος του αυτών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καθώς και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτό βεβαίως είναι προς ικανοποίηση των πολιτών. και τέλος κύριε πρόεδρε η δημιουργία ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος για τη λειτουργία και χρηματοδότηση των κομμάτων είναι πράξη βαθιά δημοκρατική. χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό χώρο ενεργών πολιτικών κομμάτων που θα φέρουν τους πολίτες στο επίκεντρο της ένωσης και θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή τους ζωή. αυτό θα σημάνει μεγαλύτερη συμμετοχή περισσότερη δημοκρατία και σε τελευταία ανάλυση περισσότερη ευρώπη. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο την κυρία Γιαννάκου. Ε, κατόπιν του, του ολοκληρώνεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 η ώρα. Περνάμε τώρα